Welcome. Αγαπητοί βουλευτέ, καλώ ήρθατε. Παρακαλώ βάλτε τις κάρτες φοφορίας Για να ξέρουμε People πόσοι θα ψηφίσουν. Who voting for the Greens? Yes. So I hope everybody is has put his voting card into the slot. Είστε έτοιμοι για να ψηφίσετε, ελπίζω. Θα ψηφίσουμε. Ποιος θα ψηφίσει εκ μέρους των πράσινων, γιατί υπάρχει ένας παραπάνω. Μια παραπάνω κάρτα δηλαδή. Και να Okay, we are 21, 21 θα ψηφ... άτομα ψηφίζουν. Ψηφίζουμε. Την έκθεση Ροζιέρο. Ξεκινάμε. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. υιοθετείτε. Τροπολογία 2. Υπέρ κατά εποχές υιοθετείται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά εποχές υιοθετείτε. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ κατά εποχές υιοθετείτε. Ήμκο 9 υπέρ κατά, αποχές υιοθετείται. Καλτ 2 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. Συμβιβασμός 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Διαθετείτε. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Διαθετείτε. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Διαθετείτε. Συμβιβασμός 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές Υιοθετείτε. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 16 υπέρ κατά εποχές Συμβασμός 4 υπέρ κατά εποχές υιοθετείται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά εποχές Oh, sorry, sorry. Amendment 7. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Συμβασμός 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Συμβασμός 6. Υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμός 7 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 2 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε, ΙΜΚΟ 9 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται ΙΜΚΟ 9 τρίτο εδάφιο υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. ΚΑΛ 4 υπέρ κατά εποχές υιοθετείται καλτ 6 υπέρ κατά εποχές υιοθετείτε καλτ 9 υπέρ κατά εποχές υιοθετείτε είναι τα 5 υπέρ κατά εποχές υιοθετείτε καλτ 10 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε, Καλτ 12 υπέρ κατά αποχές είπ, κατά, Καλτ 14 υπέρ κατά αποχές υιοθετειτε Είναι τα 4 υπέρ κατά αποχές υιοθετειτε Καλτ 15 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε, Καλτ 16 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Κάτ 17 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Κάτ 20 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Είναι τα 1 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Είναι τα 3 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται τροπολογία 50 υπέρ κατά να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά νομίζω ότι περνάει αλλά ας δούμε We are we are voting on Amendment 50, right? Okay, is the card working now? There's one one one vote missing. We are missing one. Μας λείπει ένας και ψηφίζουμε την 50. Okay. Adopted. Adopted. Υιοθετήθηκε τελικά. Τροπολογία 51 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 8 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε ΙΜΚΟ 15 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε κάλτε 7 υπέρ κατά αποχές Είναι τα 6 υπέρ κατά αποχές Είναι τα 8 υπέρ κατά αποχές είναι τα 9 υπέρ κατά αποχές είναι τα 11 υπέρ κατά αποχές είναι τα 12 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε, τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε 27, τροπολογία 27 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε, Ήμκο 7 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε, Καλτ 11 υπέρ, κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ε, adopted in τα 7 υπέρ, προηγούμενη υιοθετήθηκε βέβαια, κατά, αποχές υιοθετήθηκε, είναι τα 10 υπέρ, κατά, αποχέ, υιοθετείται, συμβασμός το υπέρ, κατά, αποχές υιοθετήθηκε, Τροπολογία 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός. Ε, τροπολογία 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Συμβασμός 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Συμβασμός 10. Υπέρ κατά αποχές υιοθετείται συμβασμός 11 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται ΙΜΚΟ 12 υπέρ για το τμήμα 2 έτσι της 12 Ήμκο 12 τμήμα 2. Υπέρ κατά αποχέ υιοθετείται. Τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχέ υιοθετείται. 44 υπέρ κατά αποχέ υιοθετείται. 45 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. Συμβασμός 12 υπέρ κατά αποχές υιοθετήθηκε τροπολογία 46 υπέρ κατά απορρίπτεται μάλλον αποχές απορρίπτεται εντάξει να ελέγξουμε το 46 συμφωνείτε Απορρίφθηκε. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 39 υπέρ κατά αποχές διαθετείται δύο υπέρ κατά αποχές διαθετείται σοτα7, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά εποχές υιοθετείται συμβασμός 13 υπέρ κατά εποχές υιοθετείται τροπολογία 30 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται τροπολογία 52 υπέρ κατά εποχές Υιοθετείτε. Τροπολογία 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Και τώρα ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία ολόκληρη την έκθεση. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Υιοθετείτε. Συγχαρητήρια κυρία Θα Θέλετε να πάρετε το λόγο. Σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο των συναδέλφων. Ήταν ε, μεγάλη ικανοποίηση να δουλέψω πάνω σε αυτήν την έκθεση. Ευχαριστώ ιδιαίτερος την ε, ομάδα, τα μέλη της ομάδας και τη βοηθό μου, την Λοντή, η οποία έκανε τεράστια δουλειά από πίσω από τα παρασκήνια για την έκθεση αυτή. We continue, uh, Και συνεχίζουμε λοιπόν τώρα την ε, ψηφοφορία στο 14, ηλεκτρονικά παρακαλώ, με ονομαστική κλίση. Λείπει μία ψήφος, άλλη μία ψήφος. Τώρα μάλιστα. Είμαστε εντάξει. Εγκρίνεται. Η 15 με διάταση χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. We continue thereby. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Στο 22. Ανταλλαγή απόψεων. Το λόγο έχει ο κ. Άντερσον που είναι εισηγητής. sorry for a second. Μισό λεπτό λέει ο Πρόεδρος. Δεν έχει καταφάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα στην αίθουσα. Uh, since we do not... Και μια δεν έχει και δεν έχει καταφτάσει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ας συνεχίσουμε στο 18. Uh, και το λόγο έχει ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα μιλήσω βουλγαρικά σας παρακαλώ λοιπόν να βάλετε τα ακουστικά σας για να ακούσετε τη μετάφραση. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ως εισηγητής για την Επιτροπή Γιούρη για την ψηφιακή αγορά θα ήθελα να σας παρουσιάσω πώς έχει η κατάσταση. Καλώς ορίζω ιδιαίτερα τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε αφυπνισμένοι σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία μετά τη συνάντηση της 9 Ιουλίου του 2015, η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε ότι η ΙΤΡΕ και η ΙΜΚΟ θα είναι οι αρμόδιες καθήλυν επιτροπές και τη... υπό, τον κανόνα, υπό τον ε, άρθρο 55 για την ψηφιακή αγορά, ενώ η Επιτροπή δική μας με την ΑΜΠΛ, την ΚΑΛΤ και την ΛΥΜΠΕ θεωρήθηκαν συναρμόδιες με το άρθρο 44. Θα επικεντρωθώ σε θέματα που άπτονται της μεταρρυθμίσης, της ε, μελλοντική ε, νομοθετική πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ήθελε να υπάρξει κατανομή των αρμοδιοτήτων και χαίρομαι που βάσει του άρθρου 54 θεωρήθηκε και ότι και η Γιούρη είναι αρμόδια σε ό,τι αφορά το δίκαιο για τις μικρές συμβάσεις, θέματα που αφοράν, αφορούν το κοινωτικό δίκτυο. Εμείς ε, επικεντρωνόμαστε στο σημαντικό δίκαιο και στα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Η μεταρρύθμιση λοιπόν σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τις σχετικές ε, παραβιάσεις. Λοιπόν, επικεντρώνομαι στην αφαίρεση των εμποδίων στο εμπόριο και εναρμόνιση των διαδικασιών σε όλες τις επιχειρήσεις προκειμένου να προωθηθεί και η καινοτομία αλλά και η ανταγωνιστικότητα. Κατά δεύτερον, μεταρρυθμίσεις στοχευμένες για να μπορέσουν να είναι πιο φορητά τα περιεχόμενα, τα ψηφιακά Ύστερα, ο ρόλος των παρόχων ε, διαδικτύου σε σχέση με τα παράνομα περιεχόμενα που διατίθενται στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε για τέτοιου είδους περιεχόμενα και θα πρέπει να περιορίσουμε την πρόσβαση σε αυτά, καθώς και την φορητότητά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναρωτηθούμε και να σκεφτούμε θέματα εφαρμογής των πνευματικών δικαιωμάτων το νομικό περιεχόμενο είναι κάτι το οποίο θα εξετάσει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Συμπερασματικά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η πρόθεση της, Ευρωπαϊκής, της Επιτροπής μας είναι να αποσυρθεί η πρόταση για τις πωλήσει και αν αυτού να προταθεί να, να γίνει μια νέα πρόταση. Θα πρέπει να σκεφτούμε το κοινό κινητικό δίκαιο για τις πωλήσει. Υπάρχουν και άλλα επιπρόσθετα θέματα και δυστυχώς τα θέματα αυτά δεν έχουν συμπεριληφθεί στην πρόταση λόγω και χρονικών περιορισμών. Για ένα λοιπόν σημείο αυτό για την συνθήκη Μαράκες. σε ό,τι αφορά την ψηφιακή κατάσταση θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη την καλύτερη πρόσβαση στο διαδικτυακό περιεχόμενο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να προστατευτεί και η οικονομία μας αλλά και οι κοινωνίες μας. Ένα άλλο βασικό ζήτημα το οποίο θα συμπεριληφθεί είναι οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων τομέων προκειμένου να μπορέσει να είναι εύρυθμη η ψηφιακή αγορά θα πρέπει να προφυλάξουμε και την πολιτισμική μας κληρονομιά, να σκεφτούμε τι γίνεται και με τον δημιουργικό κλάδο, με τα εικαστικά. Θα πρέπει να προστατεύσουμε και τον δημιουργό, τον συγγραφέα. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διάσταση της ψηφιακής ε, οικονομίας. Όπως σας ε, ανέφερα και το θέμα της φορευτότητας, του streamlining, της ε, ευρείας πρόσβασης είναι θέματα σημαντικά. Και αυτά σχετίζονται και με τη βελτίωση των κανόνων για την ε, ηλεκτρονική κυβέρνηση, τις ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες. Κάτι άλλο που θα ήθελα να τονίσω. Η σημασία του να υπάρξει διάσταση και, κατα... και διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων των επιτροπών. Αυτές οι αρμοδιότητες είναι ορισμένες μάλιστα με τρόπο προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματική λειτουργία και συνεργασία μεταξύ των επιτροπών. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία έχει παραταθεί μέχρι την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 5 η ώρα το απόγευμα 17.00. για την Ήτρα και την ΚΑΛΤ 15 Οκτωβρίου, για την Λίμπε δεν έχει οριστεί ακόμα καταληκτική ημερομηνία. Δεν έχει οριστεί ακόμα η προθεσμία. Προσβλέπω στις προτάσεις σας και ελπίζω να είναι επικοδομητική η συνεργασία μας. Ελπίζω ότι και τον Νοέμβριο στο Στρασβούργο θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το κείμενο. Θα σας καλέσω όλους τους κοιόδες ε, συντόμους σε μια σύντομη συνάντηση, στην οποία και ελπίζω να μπορέσουμε να συζητήσουμε τα βασικά ζητήματα για ένα σχέδιο, για την καινοτομία, για ένα σχέδιο, ένα οδικό χάρτη. Και θα ήθελα ευθύ εξ αρχή να προσπαθήσουμε να αφαιρέσουμε όλα τα εμπόδια. Ευχαριστώ. Mr. Ο κ. Καβαντά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. να ευχαριστήσω τον κύριο Τζουμπάσκι για την πολύ ισορροπημένη έκθεσή του που δείχνει το πώς θα οδηγηθούμε προς μια λογική εναρμόνιση των κανόνων που αφορούν την ψηφιακή αγορά. Σημειώνω ότι θέλετε η πάροχοι πρόσβαση στο ίντερνετ να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στα παράνομα περιεχόμενα που φιλοξενούν. Δεν μπορούμε να μην καταπολεμούμε και στην ψηφιακή αγορά τις παραβάσεις, ειδικά των ε, δικαιωμάτων του δημιουργού. Η ενιαία ψηφιακή αγορά θα πρέπει να λάβει υπόψη τη σημασία των ψηφιακών έργων, γιατί έτσι λειτουργεί η ψηφιακή οικονομία, αλλά παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίσει ε, τη δίκαιη ανταμοιβή δημοσιο... των δημιουργών αυτών ούτως ώστε να έχουμε μια ε, στεναρή ψηφιακή οικονομία. Το σημείο αυτό συζητήθηκε όταν αξιολογήθηκε η έκθεση της, ε, για την εφαρμογή της ε, οδηγίας InfoSoc. Νομίζω ότι έχει νόημα να ξανατονίσουμε τη σημασία της στα πλαίσια αυτής της νομοδότησης, για την οποία ευχαριστώ τον κύριο Τζομπόφσκι. Ευχαριστώ κύριο Ράντιεφ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι. Η ψηφιακή οικονομία και οι τεχνολογίες ενημέρου, επικοινωνίας έχουν τεράστιες, τεράστιο δυναμικό. Οι δυναμικές ψηφιακές αγορές μπορούν να γεννήσουν δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο και μπορούν να δημιουργήσουν εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις απασχόλησης. Σήμερα έχουμε ποικίλου κανόνε για τι ηλεκτρονικέ επικοινωνίε και τα συμβατικά θέματα. Είναι δύσκολα να μεταφέρουμε οπτικοακουστικά προϊόντα διασυνοριακά και ψηφιακό περιεχόμενο, γιατί υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών ε, και διαφορετικό πλαίσιο. Το νομικό πλαίσιο αντιστοιχεί όλο και πιο δύσκολα στην, ε, απέναντι, με τη φρενήρη ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς. Νομίζω ότι η στρατηγική για την ψηφιακή αγορά, που είναι μια δέσμη στοχευμένων κανόνων που θα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η προστασία των καταναλωτών και οι εναρμονισμένοι κανόνες για το, τις α, συμβάσεις τις διασυνοριακές, είτε φυσικών αγαθών είτε ψηφιακού περιεχομένου, θα δώσει στους καταναλωτές πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια όταν αγοράζουν online και θα ενισχύσει το διασυνοριακό εμπόριο. Οι νομοθετικές προτάσεις που θα γίνουν, ελπίζω, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μειώσουν τις διαφορές ανάμεσα στα εθνικά νομικά καθεστώτα σε ό,τι αφορά το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, το copyright και θα έχουμε ενιαία πρόσβαση ε, στο ψηφιακό περιεχόμενο και μέσω περαιτέρω ε, μέτρων εναρμόνισης και της εναρμόνισης του Ευρωπαϊκού ε, Συμβατικού Δικαίου. Θα πρέπει επίσης τα εμπορικά μητρώα να αλληλοσυνδέονται στην Ευρώπη και με αυτόν τον τρόπο τα διάφορα εθνικά συστήματα θα λειτουργούν αμφίδρομα ούτως ώστε οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να δίνουν τα στοιχεία τους στις δημόσιες αρχές μόνο μία φορά. Αλλιώς οι κυβερνήσεις να μην μπορούν να ζητούν τις ίδιες πληροφορίες πάνω από μία φορά όταν ήδη τις έχει τουλάχιστον μία κυβέρνηση ή μία εθνική αρχή. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στις ψηφιακές υπηρεσίες και την ασφάλεια, ιδίως μέσω της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε ό,τι αφορά το ρόλο των ε, παρόχων πρόσβαση στο ίντερνετ, θα πρέπει να κάνουμε μία ανάλυση εδώ. Η, η επέκταση των υποχρεώσεών του των σε σχέση με το περιεχόμενο μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα νομικής, οικονομικής και τεχνικής φύσης. Και μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Reda. Ευχαριστούμε. Κύριε Ρέντα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την έκθεσή του και που μας έδωσε και χρόνο για να δουλέψουμε λίγο πάνω στις τροπολογίες. Νομίζω ότι είναι αρκετά περίπλοκος ο φάκελος αυτός. με τους τομείς που περιλαμβάνει για τις αποκλειστικές ε, ε, αρμοδιότητες ε, των διαφόρων επιτροπών που επικαλύπτουν η μία την άλλη για, τον, για το geo-blocking κτλ. Έχω κάποιες ιδιαίτερες ανησυχίες για ένα σημείο που αναφέρεται στο σχέδιο της νομοδότησης για την ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών ίντερνετ. Υπάρχει μια σαφής ε, αντίφαση μεταξύ των, ε, του να ζητά κανείς να υπάρχει ε, υπευθυνότητα και ουδετερότητα από την άλλη, από τους παρόχους. Σε πολλές συζητήσει που έχουμε κάνει εδώ στο Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια, ας πούμε για το πακέτο τηλεπικοινωνιών, για την σύμβαση για την άκτα, είχαμε διότι αν δώσουμε την δυνατότητα λήψη αποφάσεων για την ενομιμότητα των αποφάσεων σε ε, ιδιωτικές, σε ιδιωτικούς φορείς, τότε θα πρέπει να δούμε το θέμα πολύ πιο προσεκτικά για να δούμε ακριβώς και την νομιμότητα του περιεχομένου από τις ιδιωτικές εταιρείε. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συγκέντρωση της αγοράς ε, στα χέρια ενός ή δύο ή λίγων, εν πάση περιπτώσει, ε, σημαντικών παικτών. Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη έρευνα, πολύ μεγαλύτερη αξιολόγηση επιπτώσεων, να υπάρξει μια προσέγγιση που θα βασίζεται σε ενδείξεις για την εφαρμογή για το, του δικαίου που σχετίζεται με το ίντερνετ και βεβαίω να ληφθούν υπόψη και όλες οι διαβουλεύσεις που έχουν γίνει και από την Κομισιόν σε αυτή τη ε, διαδικασία. Καλωσορίζω τα σχόλια του εισηγητού για την ε, για τα όσα είπε για την ε, συνθήκη. Ε, και βεβαίως για το copyright βεβαίως πρέπει να δούμε τα θέματα και των οικονομικών ε, πτυχών που μπορεί ε, να υπάρχουν αλλά φυσικά και τα δικαιώματα των ατόμων για την πληροφόρηση, τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, την προστασία των δικαιωμάτων του συγγραφέα και για τη διευκόλυνση των, της διασυνορικής πρόσβασης είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη και τα δικαιώματα των ε, μειονοτήτων, είτε είναι πολιτιστικά είτε είναι γλωσσικά. Να μην τους επιβάλλουμε μόνο την, ε, ε, την, μια τιμή για την πρόσβαση στην διασυνοριακή, στο διασυνοριακό ίντερνετ, αλλά βεβαίως θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα δικαιώματά τους. Γι' αυτό είναι καλό να υπάρξει αυτή η πρωτοβουλία από την Κομισιόν για, την, για μια διαβούλευση. Επίσης, οδηγία για την ε, για τις εκπομπές είναι πολύ σημαντική. Επίσης ε, θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε πολύ καλύτερη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και η αρχή θα πρέπει να είναι ότι οι δημόσιες ε, διοικήσεις θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανείς, να δρουν όσο το δυνατόν πιο διαφανώς και οι διαδικασίες να είναι απλές για τους καταναλωτές και τα δεδομένα τους να προστατεύονται όσο το δυνατόν περισσότερο. Ευχαριστώ. Thank you as uh, Ευχαριστώ κυρία Gebhardt. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την πραγματικά πάρα πολύ καλή έκθεση και τις πολύ καλές προτάσεις τις οποίες συμπεριέλαβε σε αυτή. Νομίζω ότι εδώ συγκλίνουν οι απόψει μας ότι θα πρέπει να κάτσουμε και να κοιτάξουμε πώς η ψηφιακή αγορά πρέπει να βελτιωθεί αλλά και να πλαισιωθεί όπως πρέπει. Αυτό αποτυπώνεται, πιστεύω, εξαιρετικά στις ε, προτάσεις σας. Δύο σημεία θα ήθελα να επισημάνω. Στο σημείο 1 και στο σημείο 5 έχω να αναφέρω κάποια πράγματα. Στο 1. Συμφωνώ με την αρχή. Συμφωνώ. Ωστόσο, κάπως με προβληματίζει το τελευταίο σημείο. Ότι καλεί να γίνουν ε, να υποβάλλονται οι νέες προτάσεις σε τεστ ανταγωνιστικότητας. Δεν πιστεύω ότι αυτό φυσικά μας βρίσκει αντίθετους, αλλά στο τελευταίο ψήφισμα του Κοινοβουλίου αποφασίσαμε για την ιστορική αγορά ότι δεν επαρκεί να γίνονται τεστ ανταγωνιστικότητας, αλλά και θα πρέπει να γίνονται επιπλέον στους καταναλωτές, στους ε, ε, εργαζόμενους και στους εργοδότες ε, μελέτες αντικτύπους. Ένα πακέτο, αν θέλετε, με τεστ δεν αφορά δηλαδή μόνο το θέμα την ανταγωνιστικότητα και τις επιχειρήσεις, αλλά και ποιο είναι ο αντίκτυπος στον κόσμο γενικά. Και αυτό θα πρέπει να λεφτεί υπόψη. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να γίνει κάποια τροπολογία για να το συμπληρώσω όπως σας ανέφερα. Στο 5 τώρα. Παρατηρείται με επικριτικό πνεύμα την επιλογή της χώρας υποδοχής. Συμφωνώ. Να το εξετάσουμε με κριτικό πνεύμα και θα ήθελα να είναι και ακόμα πιο έντονη διατύπωση στην παράγραφο αυτή. Γιατί σε τελική ανάλυση το θέμα εδώ είναι τι κάνουμε με τους κανονισμούς Ρώμη 1 σε ό,τι αφορά το, την προστασία του καταναλωτή και τι γίνεται σε περίπτωση που περτερεί του κοινωτικού δικαίου. Ποιο ισχύει το δίκαιο της χώρας όπου έγινε η αγορά. Αυτό δεν είναι δυνατόν να το αμφισβητήσουμε σήμερα ή πολίτε. έτσι κι αλλιώς. Έχουν σε μεγάλο θεωρούν ότι είναι μεγάλο το κύριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα πρέπει να το αφισβητήσουμε αυτό. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι ακόμα πιο έντονη η διατύπωση. Θεωρώ ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό. Να απαντήσω και σε μία παρατήρηση που έκανε ο κ. Βράντεφ. Μιλήσατε με πριντικό τρόπο για το once only principle στο e-government, ότι δηλαδή δίνονται τα στοιχεία μία φορά μόνο στην αντίστοιχη η κρατική υπηρεσία. Καλό αυτό, αλλά συνταγματικός πώς είναι τελείως αδύνατο στη Γερμανία. Σε ό,τι αφορά δηλαδή την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών ναι, είναι παραβάση αυτό. Άρα Πώς να πούμε εμείς ότι συμφωνούμε. Η κυρία Κάλλας από την Ήτρα η το έβαλε και αυτή στην έκθεσή της το στοιχείο αυτό και το τσέκαρα και το ανέφερα σε διάφορες συζητήσεις και με δημόσιες υπηρεσίες και με πολίτες και πραγματικά ήταν κατηγορηματικό το όχι από όλους. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ συγκεκριμένα και θα ήταν αντίκτυπος ε, μιας αρχής και στα συντάγματα των διαφόρων χωρών και το θέμα της προστασίας των δεδομένων θα πρέπει να αποκτήσει υψηλότερη προτεραιότητα στο Κοινοβούλιο. Αυτό ασφαλώς θα το συμφωνήσουμε και θα το συζητήσουμε εκτενώς με τους συναδέλφους από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Κυρία Γκέριγκερ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον συνάδελφο για την γνωμοτότηση και δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που ήδη ακούσαμε από τους προηγούμενους ομιλητές. Κάποιες ερωτήσεις επιτρέψτε μου να κάνω και κάποιες ε, προτάσεις. Στο σημείο 1 αναφέρεται η άρση του φραγμού στο εμπόριο. Ωραία, το καταλαβαίνουμε αυτό. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν ίσα δικαιώματα σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά το εμπόριο. Αλλά υπάρχει ας πούμε διαφορά σε ό,τι αφορά το ύψος των τελών, σε κάποιες περιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά το private copy. Και εδώ. Και αυτό παίζει μια σημασία σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα. Υπάρχουν λοιπόν σε κάποιες περιπτώσεις τέτοια, τέτοιες επιβαρύνσεις. σε κάποια κράτη. Σε κάποια άλλα κράτη δεν υπάρχουν καν τέτοιες επιβαρύνσεις. Σε κάποιες χώρες υπάρχουν διαφορές στο ύψος των ε, επιβαρύνσεων. Και σε ό,τι αφορά του φραγμού, πιστεύω ότι θα πρέπει να το προσθέσουμε. Θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο σημείο 3 τώρα. αναφέρεται η ευθύνη, η μεγαλύτερη ευθύνη για το παράνομο περιεχόμενο. Όπως και στην ε, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων θεωρώ ότι δεν είναι σωστή αυτή η διατύπωση. Θα πρέπει, μπορούμε να λέμε μεγαλύτερη ευθύνη, πιο πολύ ευθύνη. Θα πρέπει να πούμε ακριβώς ποια ευθύνη θα πρέπει να φέρουν. Είναι πολύ γενική η διατύπωση. Προκειμένου να μπορούμε να το εφαρμόσουμε και στο μέλλον αυτή η παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών είναι παροχή υπηρεσιών στη τελική ανάλυση. όπως και για παράδειγμα στους αυτοκινητοδρόμους. Μπορεί να υπάρχει πάροχος υπηρεσιών, δηλαδή η εταιρεία που έχει φτιάξει τον αυτοκινητόδρομο, αλλά δεν φταίνεται για το τι μεταφέρουν στα φορτηγά που περνάνε. Ίσως λοιπόν κάτι παρόμοιο να ισχύει και στο διαδίκτυο. Υπάρχουν παράνομα περιεχόμενα, αλλά θα πρέπει να ορίσουμε ποιο φέρει ποια ευθύνη. Δεν φτάνει να λέμε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ευθύνη. Κάτι άλλο, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησία και ό,τι αφορά την ενιαία διαμόρφωση των εξαιρέσεων. Και εδώ υπάρχουν σοβαρέ διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και αυτό επηρεάζει και την κοινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Θα πρέπει λοιπόν βαθμία να υπάρξει μια εναρμόνιση. Σε όλες τις εξαιρέσεις όμως να υπάρξει αυτή η εναρμόνιση. Όχι βέβαια σε πράγματα που έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο εκπαίδευση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και αυτό ήταν ο τελευταίο ομιλητή για το θέμα αυτό. Ο κ. Τζαμπάσκη θέλει να πάρουν το λόγο. Ε, λοιπόν μπορούμε να επανέλθουμε στο σημείο 22, μια και ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό. Έχουμε εδώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λόγο έχει ο κύριος Άντερσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ε, συνθήκη για την ε, πρόσβαση στο δικτύο για άτομα που έχουν ειδικέ ανάγκε ή που είναι τυφλά κτλ. Και η επικύρωσή της ε, έχει περάσει από όλα τα θεσμικά όργανα και έχει συζητηθεί εδώ και πολύ καιρό. Πολλές άλλες χώρες την έχουν επικυρώσει και σύντομα μάλλον θα τεθεί και σε ισχύ. Ε, η δική μου εντύπωση είναι ότι υπάρχει μεγάλη ισχυρή στήριξη εντός του Κοινοβουλίου για το ότι όντως θα πρέπει να επικυρωθεί, αλλά το θέμα μάλλον κολλάει στο Συμβούλιο. Η Κομισιόν έχει προτείνει σύντομη, άμεση επικύρωση και έχουν υπάρξει και κάποιες τελευταίες εξελίξεις όπου η Κομισιόν ε, έχει προετοιμαστεί να πάει στο δικαστήριο με το θέμα αυτό. Ε, είναι λυπηρό, αλλά η Κομισιόν πρέπει να το κάνει αυτό. Νομίζω ότι είναι σωστός ο τρόπος που θα ακολουθήσει και θα ήθελα φυσικά να ακούσουμε περισσότερο από την Κομισιόν για το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, may I ask Mrs. Ευχαριστώ. Η κυρία Πράτ, παρακαλώ να πάρει το λόγο. Ε, thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Άντερσον που μας υπενθύμησε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα σχετικά με την επικύρωση της συνθήκης του Μαρακές. Όπως είπε ο εισηγητής, η Κομισιόν ήδη έχει υποβάλει στο Συμβούλιο το θέμα αυτό της, κοινο... της επικύρωσης της σύμβασης η οποία ήδη έχει υπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έθεσε ε, λοιπόν το θέμα αυτό εδώ και πολύ καιρό στο Συμβούλιο, μάλιστα συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, δηλαδή περίπου ένα χρόνο πριν. Η πρόταση της Κομισιόν για την επικύρωση της συνθήκης βασίζεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. Αυτή είναι η άποψη της Κομισιόν και της Ζωμικής Υπηρεσίας. Ε, δεν, δεν υπάρχει αντίρρηση από την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου και βασίζεται στην άποψη ότι τα δικαιώματα που πλήττονται από την ε, υποχρεωτική εξαίρεση από την συνθήκη του Μαρακές για, τους, ε, για τα άτομα που έχουν κάποιες αναπηρίες έχουν εναρμονιστεί αυτά τα δικαιώματα ε, πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ε, οδηγίας Συμφωσόκ του 2011. Επίσης η συνθήκη προβλέπει ε, κάποια, κάποια, κάποιες ε, αλλαγές για τα προσβάσιμα έγγραφα για τα άτομα αυτά με αναπηρία και μάλιστα έχουν υπάρξει και αρκετές αποφάσεις του δικαστηρίου που επιβεβαιώνουν την αρμοδιότητα της Ένωσης ε, επ' αυτού. Γι' αυτό η Κομισιόν θεωρεί ότι το θέμα εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης και αυτό επιτρέπει να υπάρξει μία επικύρωση για την συνθήκη η οποία βεβαίως θα είναι δεσμευτική για τα 28 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι έχει γίνει τώρα μετά, από τότε που ε, τέθησε το τραπέζι του Συμβουλίου η πρόταση. Ε, ήμασταν προς το τέλος του 2014 έγιναν συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και μετά, κατά τη διάρκεια της Λετωνική Προεδρία, όπου πήγε το θέμα στην Κορεπέρ, γιατί ήταν απολύτω σαφέ ότι το θέμα δεν ήταν τελικά τεχνικό, δεν ήταν καν άμεσα σχετιζόμενο με την συνθήκη του Μαρακές. Ήταν οριζόντιο θέμα της ε, αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι υπήρχε μια ασυμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Έγιναν αρκετές ανταλλαγές απόψεων σε επίπεδο Κορεπέρ για να ε, καταλήξουμε τελικά σε ένα συμβασμό, σε μια συμβαστική λύση. Ε, η Κομισιόν έδειξε μεγάλη ευελιξία, προσπάθησε να δώσει πολλές εναλλακτικέ, ε, μάλιστα έβαλε πολύ φαντασία σε μερικές, έτσι ώστε να ξεμπλοκάρει η υπόθεση και να γίνει η επικύρωση της συνθήκης. Τελευταία φορά που συζητήθηκε το θέμα αυτό στην Κορεπέρ ήταν στις 6 Μαΐου του 2015. Σε εκείνη τη φάση κατέστη πλέον σαφές ότι βρισκόμασταν σε αδιέξοδο. Έχουμε μια πολύ σημαντική πλειοψηφία, αλλά όχι επαρκή κρατών μελών που σκέφτονται να συμφωνήσουν με την πρόταση και τη συμβαστική λύση που υπάρχει ε, το γεγονό ότι είμαστε στα πλαίσια τη αποκλειστική αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση μα διευκολύνει μεν, αλλά δεν έχουμε την απαραίτητη στήριξη των, ε, του απαραίτητου αριθμού μάλλον κρατών μελών για να προχωρήσουμε με την επικύρωση. ώστε να πάει μετά στο, να αποσταλεί στο Κοινοβούλιο. Και λόγω αυτού λοιπόν του αδιεξόδου στο οποίο βρισκόμαστε και για να μην χάσουμε άλλο χρόνο, η Κομισιόν αποφάσισε να ζητήσει γνωμοδότηση του δικαστηρίου Οπότε η Κομισιόν έχει ζητήσει από το δικαστήριο να λάβει θέση για το αν η συνθήκη του Μαρακές και η επικύρωσή της εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης ή αν είναι ε, αρμοδιότητα κρατών μελών. Αυτή η γνωμοδότηση, ε, μάλλον το αίτημα για τη γνωμοδότηση αιστάλλει στο δικαστήριο 17 Ιουλίου με αριθμό 315 είναι δημόσια προσβάσιμο το έγγραφο. Ε, λυπάται η Κομισιόν που έφτασε στο σημείο αυτό η κατάσταση, αλλά δεν θέλαμε να χάσουμε άλλο χρόνο. Η πρότασή μας για την επικύρωση της συνθήκης βεβαίως εξακολουθεί να υπάρχει. Ε, είναι ακόμα στα χέρια του Συμβουλίου το, αν το Συμβούλιο θέλει να αποφασίσει ότι θέλει να προχωρήσει και να βρει μια λύση και να επικυρώσει το, τη συνθήκη, μπορεί ακόμη να γίνει αυτό. Απλώς εμείς δεν θέλουμε να μπλοκαριστεί τελείως η ε, κατάσταση και να μην να σταματήσει να γίνεται το οτιδήποτε. Ήταν σαφές πριν το καλοκαίρι ότι υπήρχε αυτός ο κίνδυνος. Απολύτου δηλαδή... Ε, απόλυτη στασιμότητα. Αυτά, Πρόεδρε, από μένα. Αν υπάρχουν ερωτήματα, ευχαριστώ να απαντήσω. Thank you very much. Ε, Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκασπαρό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που ε, θέσατε το θέμα για τη συνθήκη του Μαρακές ε, στην ημερήσια διάταξη και ευχαριστώ και τον κύριο Άντερσον. Νομίζω ότι ε, έχουμε έτσι μια γενική εικόνα της κατάστασης δεδομένου του ότι το Κοινοβούλιο το έχει πει συχνά. Και όπως ε, υπενθύμισε και ο κύριος Άντερσον, από τις 29 Απριλίου συνέβησαν διάφορα πράγματα, όπου στην ε, Ολομέλεια στο Στρασβούργο, στη συνεδρίαση στο Στρασβούργο, είχαμε την έκφραση της στήριξης της Κομισιόν. Η Ισπανία ε, επικύρωσε επίσης την συμφωνία του Μαρακές, αλλά η σύμβαση για το ε, δικαίωμα των ε, αναπήρων ε, αναγνώρισε ότι υπάρχει μια απίστευτη ότι, υπάρχει, ότι είναι προτεραιότητα και ότι τώρα εμείς το τι έχουμε κάνει. Θα πρέπει να ξαναζητήσουμε, να ξαναπευθυνθούμε στο Συμβούλιο και νομίζω ότι είναι χρήσιμη, ε, χρήσιμο το αίτημα για γνωμοδότηση του δικαστηρίου αλλά φοβάμαι, και ας μου πει η Κομισιόν, ότι θα υπάρχει ένα πρόβλημα χρονικό για να πάρουμε απάντηση από το δικαστήριο. Γιατί. Έχω την αίσθηση ότι γίνεται μία απόπειρα εδώ πέρα. Ε, εδώ ο συγγητής βέβαια σε σχέση με το copyright ε, μου είπε ότι, είπε ότι η οδηγία 29 σε σχέση με τη συμφωνία του Μαρακές πρέπει να ακολουθήσει διαφορετική πορεία. Και δεν θα ήθελα λοιπόν η περίπλοκη αυτή η κατάσταση αδιεξόδου ε, στην οποία περιήλθε η συμφωνία του Μαρακές να συμπεριλάβει και την οδηγία 29 που αφορά τους κανόνες για το copyright. Είναι κρίμα, δεν το θεωρώ σωστό σε σχέση με τις δεσμεύσει που η συμφωνία του Μαρακές ε, έχει αναλάβει και για τα δικαιώματα τα οποία θέλουμε να προστατεύσουμε. Ευχαριστώ. Thank you very much. Before Εγώ ευχαριστώ. Να πω ότι το Συμβούλιο μπορεί να προχωρήσει με την επικύρωση. Η Κομισιόν έχει ζητήσει με την γνωμοδότηση του, του δικαστηρίου, το είπε η κυρία Πράτη πολύ έντονα, το Συμβούλιο όμως μπορεί να προχωρήσει αν θέλει στην επικύρωση, το είπαμε και πριν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το θέμα που δείξατε μόλις είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Το γεγονό ότι η Κομισιόν τώρα ζητά την βοήθεια του δικαστηρίου. Από τη μια δεν θα πρέπει να σταματήσει τη δουλειά που ε, έχει υποσχεθεί ε, ο πρόεδρος ε, της Κομισιόν να γίνει επ' αυτού. Αυτό θα πρέπει να γίνει, να συνεχίσουν δηλαδή οι εργασίες, όσο το δικαστήριο θα ε, εκπονεί την γνωμοδότησή του. Και νομίζω ότι το έχουμε... Έχει ξαναϋποθεί αυτό. Και έχει υπάρξει έτσι μια απορία γιατί υπάρχει τέτοιο θέμα αποκλειστική ή μη αρμοδιότητα Ευρωπαϊκή Ένωση, μια που η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει νομοθετήσει ευρέω τον τομέα αυτό. Ίσως αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει μια εξαίρεση για τα άτομα με αναπηρία και υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις για το copyright, ήδη υποχρεωτικέ και ήδη εφαρμοστές. Να ευχαριστήσω την Κομισιόν που προσπάθησε να βρει μια λύση και να τονίσω ότι όντως αυτό το θέμα είναι θέμα προστασίας θεμελιδών δικαιωμάτων. Άτομα που έχουν ε, προβλήματα όρασης, ε, δεν μπορούν να εξασκήσουν τα ε, δικαιώματα της εκπαίδευσης ε, ή της άμεσης πρόσβασης σε οτιδήποτε και αυτό νομίζω ότι πρέπει άμεσα να διορθωθεί. Ευχαριστώ. Κυρία, κυρία Χάνιμπαλ, συμφωνώ απόλυτα με όλα όσα έχουν υποθεί. Νομίζω ότι είναι φρικόδες αυτό που συμβαίνει. Επι... Εδώ θέλουμε να επιτρέψουμε σε ανθρώπους να κάνουν αυτό που εμείς χωρίς κανένα πρόβλημα και χαλαρά κάνουμε. Είναι κρίμα, είναι φρικτό που καθυστερείται τόσο αυτό το θέμα. Και θέλω να ευχαριστήσω και την Κομισιόν για τη δουλειά που έκανε σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε κάτι ως Επιτροπή, εμείς, Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι να μάθει το Συμβούλιο την άποψη τη δική μας και άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών που εμπλέκονται, ούτω ώστε να επικυρωθεί αυτή η συμφωνία. Και τα άτομα τα οποία έχουν προβλήματα όρασης να αποκτήσουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους εξημών. Με ενημέρωσαν ότι χθε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου αποφάσισε να υποβάλουμε παρατηρήσεις στα πλαίσια της διαδικασίας νομοδότησης. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν. Η κυρία Άντερσον θέλει να ξαναπάρει το λόγο. Ο κύριος Άντερσον. Εν συνεχεία, μια άλλη ερώτηση. Εάν ε, το δικαστήριο δώσει με τη γνωμοδότησή του και όλοι θεωρούμε ότι θα πει ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το Συμβούλιο θα, συμμορφωθεί με τη γνωμοδότηση αυτή του δικαστηρίου. Γιατί πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι κάνει το Συμβούλιο. Ο τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρει το Συμβούλιο αρχίζει να γίνεται όνειδος. Και εγώ διαρωτώ μου θα τόλμα και κανένας ή θα ήθελε κανένας να θέσει αυτό το ερώτημα. ότι με αυτά τελειώσαμε τη σημερινή συζήτηση για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ και συνεχίζουμε με το σημείο 19. Σχέδιο γνωμοδότησης, υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στο χώρο της φορολογίας. Ο κ. Τζαμπάσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Όσο εισηγητής της Γιούρη για την προτινόμενη οδηγία για την τροποποίηση της 2011 ε, 16 για την αυτόματη υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών στο τομέα της φορολογίας, έχω υποβάλει διάφορες τροπολογίες και ελπίζω οι συνάδελφοι της ΕΚΟΝ να τις λάβουν υπόψη. Ε, προ, προτείνοντας τις τροπολογίες μου, προσπάθησα να μην ξεπεράσω τα όρια της εντολής της Γιούρη, γιατί υπάρχει και η ειδική επιτροπή της ΙΤΑΞΑ. Ε, ε, που μπορεί να προτείνει διάφορα μέτρα και δεν θέλω να υπάρξουν επικαλύψεις. Ελπίζω ότι οι συνάδελφοι θα με βοηθήσουν για να παραμείνουμε στα πλαίσια της εντολής μας και να κάνουμε τροπολογίες μόνο μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το πλαίσιο της Γιούρη. Και αν θέλετε να υποβάλλετε τροπολογίες ε, για άλλα τμήματα της προτινόμενης ε, οδηγίας, παρακαλώ να τις υποβάλλετε μέσω των συναδέλφων της ΕΚΟΝ. Ε, θα είμαι σύντομο και ελπίζω να έχουμε μια επικοδομητική συζήτηση με τους σκιώδεις εισηγητές. Γενικά υποστηρίζω την ε, προτινόμενη τροπολογία της οδηγίας. Ε, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να προστατεύονται τα εμπιστευτικά στοιχεία των φορολογουμένων. Επίσης θα πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο το διοικητικό άχθος. Επομένως θα πρέπει να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση και θα πρέπει τα υποβαλλόμενα ε, στοιχεία να εξυπηρετούν το στόχο της οδηγίας. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να συζητήσουμε τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό ή ε, επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό. Ε, το να μπουν σε ένα νομικό κείμενο όταν δεν έχουν αναλυθεί αρκετά, νομίζω ότι θα επηρεάσει αρνητικά την προτινόμενη τροποποίηση της ε, οδηγίας, διότι θα οδηγήσει σε νομικά παραθυράκια και δεν θα μας επιτρέψει την άνετη εφαρμογή της προτινόμενης ε, νομοθεσίας. Θα ήθελα να παραθέσω την γνωμοδότηση του Σουηδικού Κοινοβουλίου που υποβλήθηκε ε, με βάση το άρθρο 16 του πρωτοκόλλου 22 της, λειτουργίας, της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοβούλιο της Σουηδίας ε, εδώ παραβιάζεται από κάποιες έννοιες η αρχή της ε, επικουρικότητας. Η Κομισιόν προτείνει να... Ή μάλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να σας πω ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί εθνική φορολογική αρχή. Το θέμα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και θα ήθελα η σχετική παράθεση να διαγραφεί. Θα πρέπει οι φορολογικέ αρχέ να συνεργάζονται μεταξύ του, να ανταλλάσσουν πληροφορίε μεταξύ του. Αλλά αυτέ οι πληροφορίε μπορεί να αναλυθούν μόνο από αρμόδιε αρχέ που υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες ε, επιστατικότητας με βάση το άρθρο 3 της τη οδηγία. Επίσης, η γνωμοδότηση Τη Ευρωπαϊκή Αρχής Προστασία των Δεδομένων ε, πηγαίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Η ανταλλαγή πληροφοριών, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν. Αλλά οποτεδήποτε προβλέπονται προθεσμίες, θα πρέπει να είναι λογικές προθεσμίες. Θα πρέπει να μπορούμε να τις στηρίσουμε στην πράξη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αναδρομικότητα και την ανδρομική ανταλλαγή, ανταλλαγή πληροφοριών. Η δεκαετία είναι τεράστια χρονική διάρκεια και θα πρότεινα την πενταετία. Σε ό,τι αφορά τη θέση σε ισχύ τη προτινόμενη ε, τροποποίηση οδηγία, τη αλλαγή τη νέα οδηγία, τα κράτη-μέλη, με βάση την πρόταση, θα έχουν από τις 31 Δεκεμβρίου του 2015 ως ε, προθεσμία για να τροποποιήσουν την ε, νομοθεσία τους και θα πρέπει να ξεκινήσουν την εφαρμογή της νέας οδηγίας από 1η Πρώτου 2016. Είναι πολύ σύντομη, πολύ σφιχτή η προθεσμία που θα επιβαρύνει τα μάλα τις εθνικές φορολογικές αρχές. Η νέα οδηγία, η τροποποιημένη, θα πρέπει να εφαρμοστεί 12 μήνες μετά τη θέση σε ισχύ, κατά την απόψή μου. Είναι λογικό να δώσουμε στα κράτη-μέλη παρκές χρονικό διάστημα για να αλλάξουν τις νομοθεσίες τους. Θα ήθελα να ακούσω τώρα τι άποψη έχουν οι σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ για την προσοχή. Ε, ε, Σας ευχαριστώ και πρωτού δώσω το λόγο στον κύριο Κέστερ. Θα ήθελα να πω ότι δεν ξέρω κατά πόσον τονίσατε ότι η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες είναι 22 Σεπτεμβρίου. 22. Μικρής Κέστερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι η έκθεση δεν ε, επαρκεί για τις ε, απαιτήσει και τις προδιαγραφές για την φορολογική πολιτική μετά το LuxLeaks. Είναι θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος η φορολογική πολιτική και η αντίληψη του κοινού για την φορολογική πολιτική είναι καθοριστική και για τις εξελίξεις σε σχέση με την αποδοχή ή μη της Ευρώπης. Και άρα πιστεύω ότι θα πρέπει να το γεγονός ότι είναι ένα δισεκατομμύριο χάνεται λόγω φοροαποφυγής από τα κράτη-μέλη είναι σκάνδαλο και θα πρέπει να είμαστε πιο σαφείς λοιπόν από αυτά που προτείνονται στις ε, προτάσεις. Επιπρόσθετα, στις δημόσιες υπηρεσίες αντιμετωπίσουμε και φτώχεια του κράτους, ε, ανεπάρκεια σε ό,τι αφορά τη συντήρηση των υποδομών, για παράδειγμα. Και αυτό καθιστά σαφές ε, το πόσο σημαντική είναι η σωστή φορολογική πολιτική, μια σωστή ευρωπαϊκή φορολογική πολιτική, η οποία θα οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου θα συνεισφέρουν τα όσα αναλογούν οι μεγάλες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα με τα κύματα των προσφύγων. Εδώ θα πρέπει να διαθέσουμε επιπρόσθετους πόρους. Προκειμένου να υπάρχει σωστή χρηματοδότηση χρειάζεται και μια σωστή τοποθέτηση. Και οι τροπολογίες ακολουθούν πιο μετριοπαθή προσέγγιση. Εγώ πιστεύω ότι η φοροαποφυγή, η φορολογική παράδειση θα πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστούν με επιθετικό τρόπο. Και είναι σωστό το γεγονός ότι μιλάμε για έναν επιθετικό τρόπο αντιμετώπισης και αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί. Δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να συμπεριλάβουμε ελαφριά διατυπώσεις και η μείωση του χρονικού ορίου σε πέντε έτη θεωρούμε ότι από πλευρά των σοσιαλδημοκρατών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Θα θέλαμε λοιπόν να εκφράσουμε την ένστασή μας εδώ. Και πιστεύω επίσης ότι οι προθεσμίες όπως προβλέπονται είναι σωστές και λογικές και δεν έχει νόημα να βελτιώσουμε τις προθεσμίες αυτές. Δεν θα μας βοηθήσει αυτό να καταρτήσουμε μια σωστή φορολογική πολιτική. Θα πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στην Ευρώπη ότι χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες και θα πρέπει να σταματήσουμε τις ασάφειες οι οποίες επιτρέπουν σε τελική ανάλυση την φοροδιαφυγή, την φοροαποφυγή και για το μέλλον. Ευχαριστώ. Κύριος Ντιουράν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν πολύ, διατυπώθηκε με πολύ εύγλωτο τρόπο, δεν θα το επαναλάβω, γιατί συμφωνώ απόλυτα. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για τη δουλειά του. Νομίζω ότι το θέμα που τίθεται τώρα είναι να δούμε εάν θέλουμε να διατηρήσουμε ε, τον φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν αντίθετα θα προσπαθήσουμε να πάμε προς μια λογική αποφυγής αυτού του φορολογικού ανταγωνισμού. Γιατί ο ανταγωνισμός μεταξύ των ε, κρατών ε, οδηγεί σε dumping, σε φορολογικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάποια κράτη-μέλη και σε, σε μείωση των φορολογικών εσόδων. Έτσι. Το ερώτημα που θέτει η γνωμοδότησή σας είναι ξεκάθαρο, είναι τι Ευρώπη θέλουμε. Και δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη συζήτηση αυτή, παρότι δεν θα την κάνουμε στα πλαίσια αυτή της οδηγίας και δεν θα, τη ρυθμίσουμε, ναι, θα το ρυθμίσουμε το θέμα εδώ. Ίσως πρέπει να πάμε στη γνωμοδότησή σα λίγο πιο μακριά. Ίσως θα πρέπει τα πράγματα να ξεκαθαριστούν οριστικά. Από τη μία έχουμε την άποψη της Κομισιόν και αυτή την οδηγία ε, που συμμερίζεται και ο Γιούνκερ στις παρεμβάσεις του. Δηλαδή ό,τι συνέβη στο παρελθόν που θα πρέπει να σταματήσει. Τα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, ειδικά στους προπολογισμούς διαφόρων ε, κρατών και θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια σύγκλησης. Είναι πολιτική επιλογή. Μπορούμε να κάνουμε άλλες επιλογές, της επικουρικότητας, της, ε, μια εθνική επιλογή, ε, ο κάθε ένας να φορολογεί ό,τι θέλει, αλλά αυτό που είναι επικίνδυνο, εντάξει, ίσως είναι λίγο υπερβολικό όρο, αλλά τουλάχιστον δύσκολο, είναι να μείνουμε στη μέση και να πούμε ούτε έτσι ούτε αλλιώ. Ας πούμε ότι θέλουμε τη σύγκληση. Αυτό λέει η οδηγία, αν το θέλουμε. Αλλά αν, διαγράψουμε τους όρους αυτούς που θέλετε να διαγράψετε, ε, είναι σαν να λέτε θέλουμε να μείνουμε σε αυτή τη λογική. Εγώ συμφωνώ με την ε, έκθεση, ε, και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε μια πραγματική συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Θέλουμε περισσότερο φορολογική ομοιομορφία ή θέλουμε περισσότερη επικουρικότητα. Ε, το θέσατε, ίσως όχι επαρκώς. Πάντως σας ευχαριστώ που δώσατε τη γνώμη σας. Και εγώ σας λέω τη δική μου ξεκάθαρα. Ήταν ο τελευταίος ο μιλητής, ο κύριος Τζαμπάσκι. Θέλει να συνοψίσει. Ευχαριστώ χωρίς μικρόφωνο, ο μιλητής. края на краищата това изблъсъки на а, идеи. Така че благодаря за мненията ви. Σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ επικοδομητικό. Κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τι ε, απόψει σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούμε και την κριτική. Έχω μια πολιτική τοποθέτηση και θέση και σε κάποιε περιπτώσει θα πρέπει να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, πολύ φοβάμαι. Σε ό,τι αφορά τι προθεσμίε, σε κάποια κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένως και τη Βουλγαρία, οι προθεσμίε που προβλέπει και ο ποινικό κώδικα είναι πενταετής. Δεν μπορεί κανείς να κάνει έρευνα αναδρομικά μετά από 10 χρόνια. Και είτε θα κληθούμε να αλλάξουμε όλο το ευρωπαϊκό, την ευρωπαϊκή νομοθεσία, είτε θα πρέπει να συμφωνούμε, να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Γι' αυτό λοιπόν πρότεινα την πενταετία αυτή προθεσμία. Θα συζητήσουμε το θέμα όμως αυτό σε διάφορες περιστάσεις στο μέλλον Προσβλέπω στις απόψεις σας και με χαρά θα απαντήσω. Uh, thank you. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και έτσι ολοκληρώσαμε και το σημείο 19 και έχουμε το 20 στην ατζέντα. Έχουμε τον έλεγχο τριών ε, μέτρο πράξεων κάθε εξουσιοδότηση. Δεν έχουμε τον κύριο Χρυσόγωνο εδώ πέρα μαζί μας σήμερα. Ο εισηγητής θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε ένσταση κατά των προτινόμενων μέτρων. Είχατε εδώ την ευκαιρία να διαβάσετε τα προτινόμενα μέτρα. Έχετε αντιρρήσεις, σχόλια παρακαλώ, ως προς αυτό. Όχι. Πριν ολοκληρώσουμε λοιπόν την πρωινή. Πριν ολοκληρώσουμε την πρωινή συνεδρίαση, θα ήθελα να σας διαβάσω τις αποφάσεις των συντονιστών που ελήφθησαν σήμερα το πρωί. Καταρχάς, ό,τι αφορά τον ορισμό εισηγητών. για την παρακολούθηση της εφαρμογής ε, ε, του κοινωνικού δικαίου για το 2014 στους πράσινους, ε, δεν έχει ακόμα οριστεί το ποιος, εφαρμογή του κανονισμού 1049-2001 προς την κυρία Χάουταλα, εκπροσώπηση των οργαζομένων σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων στην Ευρώπη, στον κύριο Κάσπαρα καταλληλότητα του νομοθετικού πλαισίου για τους καταναλωτές σε ό,τι αφορά την ψηφιακή ε, σφαίρα προς τον κύριο Κάριμ. Και έχουμε με πέντε υποθέσεις ασυλίας, Ιστβαν Ουιχελ, ο κύριος Βιέσκα, για τον Γεώργιο Κίρτσο, η κυρία Ρέγνερ, για τον κύριο Στέλιο Κούλογλου, εγώ ο ίδιος προσωπικά, για τον κύριο Σεκέρισκη, η κυρία Χάουταλα και για τον Ρόμπερτ Ιβασκίεβιτς, ο κύριος Χρυσόγονος. Στη συνέχεια οι συντονιστές αποφάσισαν να ζητήσουν ε, διεξαγωγή μελέτη για την πρόληψη ε, εμπορίου και σε αλληλετημένες πολιτισμικές περιοχές. Αποφασίσαμε επίσης να ακυρώσουμε την συνεδρίαση της ε, Επιτροπής στις 21-22 Δεκεμβρίου 2015 και να την αντικαταστήσουμε μία συνάντηση στις Βρυξέλλες στις 11 Ιανουαρίου του 2016. Μία συνάντηση στο Στρασβούργο θα λάβει, θα λάβει χώρα στις 14 ε, Δεκεμβρίου φέτος το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εγκρίθηκε για το 2016 και στη συνέχεια οι συντονιστές ορίζουσαν την κυρία Κομοντίνη και την κυρία Ροζιέρ στην αντιπροσωπεία για τη συνάντηση IGF το Νοέμβριο του 2015. Οι συντονιστές αποφάσισαν να καλέσουν την Επιτροπή Γεωργίευα και το Γενικό Γραμματέρα Ιταλιέλες για μια ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το διοικητικό δίκαιο, σε ό,τι αφορά ε, μάλλον μια μελλοντική συνάντηση της Επιτροπής. Επίσης, οι συντονιστές αποφάσισαν να διοργανώσουν ακρόαση για την διαθεσμική συμφωνία, για την καλύτερη ε, νομοθεσία, στην οποία θα συμπεριληφθεί και ο κ. Τίμερμαντς και ο κ. Βαρχόφστατ και επιπρόσθετα να προβλεφθεί και συζήτηση για το πώς έχουν οι διαπραγματεύσει και πώς εκτιλήσονται. Οι συντονιστές ενέκριναν το σχέδιο ημερήσιας διάταξης για την ακρόαση του Νοεμβρίου, για την μεταρρύθμιση του κανονισμού Βρυξέλλες 2 και οι, οι, οι συντονιστές συμφώνησαν να επανεποβάλλουν την πρόταση για τη θερινή ώρα που είχε υποβληθεί το Μάιο του 2015 και τέλος ε, ορίσαμε την κυρία Αντελβο ως προσωρινή εισηγήτρια για τη μεταρρύθμιση του δικαστηρίου ε, μιας και απουσιάζει ο κύριος Μερινού Αντίτου. Αυτές οι αποφάσεις των συντονιστών. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη συμμετοχή σας στην πρωινή συνεδρίαση. Τα λέμε στις 3. Και καλή όρεξη.